Cari colleghi, la seduta è ripresa. Ε, επανάληψη τη συνεδρίαση. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτο σημείο τη σημερινή διάταξη. προβλέπει την δήλωση του Συμβουλίου εξ ονόματο του Αντιπροέδρου της Επιτροπή, είπα τη εκπροσώπου για τι εξωτερικέ υποθέσει και την πολιτική ασφάλεια για την Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινή. Πριν να δώσω το λόγο στον κύριο Καστέλ, θα σας διαβάσω ένα απόκομμα επιστολής που, είναι, που απευθύνεται στους ευρωβουλευτές από τους ε, γιους της Σακινέ ακριβώς για την ε, συζήτηση για την Παγκόσμια ημέρα κατά τη θανατικής ποινής. Σας ευχαριστούμε για την δέσμευσή σας και την προσοχή σας, την οποία δείξατε ε, για την μητέρα μας σε η μόνη μας ελπίδα είναι η διεθνή κοινότητα και γι' αυτό το λόγο ζητάμε από το Ευρωκοινοβούλιο να παρέμβει με αποφασιστικό τρόπο με κάθε μέσο που έχει στη διαθέσή του. Ε, ώστε να βοηθήσει τη μητέρα μας και σας γετεύουμε να μην εγκαταλείψετε και να δεχτείτε αυτό το αίτημα βοήθειας ώστε, ώστε τέτοιου είδους πρωτόγονες ε, ε, τιμωρίες όπως ο λιθοβολισμός να απαγορευτούν για πάντα. Σας χαιρετούμε. Παρακαλώ, ο κύριος Καστέλ έχει το λόγο. Merci, Madame σας ευχαριστώ. Ε, Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Πρόεδρος μόλις τον έφερε ε, στο όνομα της είπα της εκπροσώπου Λέδης Άστον παίρνω το λόγο για αυτή την παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής. Όπως γνωρίζετε η θανατική ποινή, η εφαρμογή μάλλον της θανατικής ποινής σε ολόκληρο τον κόσμο παρουσιάζει αντιφατική εικόνα. Από τη μια πλευρά τα περισσότερα κράτη έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή είτε μέσω της νομοθεσίας τους είτε στην πράξη μόνο. Και ο αριθμός των κρατών που καταργούν τη θενατική ποινή αυξάνεται διαρκώς. Αυτό βλέπουμε να περιορίζεται λοιπόν σε όλες τις χώρες. Από την άλλη πλευρά, ο αριθμός και ο τρόπος εφαρμογής της θανατικής ποινής σε ολόκληρο τον κόσμο Δυστυχώ ε, παραμένει ανησυχητικό. 5.679 ε, ε, εκτελέσεις το 2009. Είναι δηλαδή 5.679 ε, εκτελέσεις ε, παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Και Άρα η δουλειά μας ε, πόρο απέχει από το τέλος της. Ε, επιπλέον γνωρίζουμε όλοι ότι εκεί όπου η θανατική ποινή παραμένει ενισχύει υπάρχουν και σοβαρά προβλήματα όπως ο σεβασμός των προτύπων και των διεθνών ε, προδιαγραφών για την εφαρμογή της θανατικής ποινής στα πιο σοβαρά εγκλήματα. Ο αποκλεισμό των προθεσμιών, η εγγύηση μιας ε, Δίκη Σε Το συμπέρασμα στα θέματα αυτά είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει χώρο για ε, αυταρέσκεια. Και γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όποια μέσα έχουμε στη διαθέσή μα τη διπλωματική οδό, την ευαισθητοποίηση του κοινού, για την υλοποίηση των του στόχου μας και γι' αυτό η ως εκπρόσωπος έχει καταστήσει την δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάργηση της θανατικής ποινής προσωπική της υπόθεση. Και τι σημαίνει όμως κάτι τέτοιο συγκεκριμένα. Η μελλοντική υπηρεσία, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση θα μπορεί να στηριχθεί στο γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη είναι σήμερα ο πρώτο θεσμικό φορέα που στηρίζει τον αγώνα κατά τη θανατική ποινή, αλλά η υπηρεσία θα αντιπροσωπεύσει επίση και θα είναι και η ευκαιρία να ε, αξιοποιήσουμε καλύτερα το δικό μας δυναμικό. Θα ενισχύσει τις δυνατότητές μας να μιλήσουμε με μια φωνή μόνο. Και αυτό θα μας δώσει την ευκαιρία να κινητοποιήσουμε καλύτερα και να διασυνδέσουμε καλύτερα όλα τα διαθέσιμα μέσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην καταπολέμηση της θενατικής ποινής. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεντρώνει τις δυνάμεις της και τις ενώνει με άλλους διεθνείς οργανισμούς και πολυμερείς δραστήριους οργανισμούς στην προώθηση της κατάργησης της θανατικής ποινής. Το ψήφισμα και το μορατόριο για την προσφυγή στη θανατική ποινή που προβλέπεται από την 65η συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τώρα το φέτος το φθινόπωρο θα πρέπει να δώσει, ανοίξει το δρόμο για μια καθολική κατάργηση της θανατικής ποινή. Θέλουμε να διευρύνουμε την τάση προς την κατάργηση που διαπιστώνεται σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Η στενή συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένα ακόμη ατού στον αγώνα κατά της θανατικής ποινή. Ω προς αυτό και πολύ συγκεκριμένα θα ενώσουμε τις προσπάθειές μας για παράδειγμα για να ενθαρρύνουμε τη Λευκορωσία να καταργήσει τη θανατική ποινή ιδιαίτερα με την διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων στο ΜΙΣ κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας ημέρας. Καθώς πιστεύουμε πως η κατάρριση θανατικής ποινής είναι βασική προϋπόθεση για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων είμαστε αντίθετη της επιβολής της σε κάθε περίπτωση και υπό οποιασδήποτε συνθήκες και είμαστε έτοιμοι να καλέσουμε για την καθολική της κατάργηση που παραμένει στόχος μας βασικός για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και επιβεβαιώνω εδώ εκ μέρου τη Λέδη Άστον την βούλησή μα και την αποφασιστικότητά μα η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την παγκόσμια κατάργηση θανατική πηγή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να διευκρινίσω ότι κατόπιν προτάσεω τη διασκέψη των Πρόεδρων θα γίνει συζήτηση με ένα μόνο βουλευτή εκ μέρους κάθε πολιτικής ομάδας. Και ως εκ τούτου δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία του ΚΑΤΣΤΙΑΗ. Ξεκινούμε με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τον κύριο Κούκαν για δύο λεπτά. Thank you very much, Madam Chair. This... Στο πολύ κυρία Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε αξίες και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πρέπει να τα προστατεύουμε παγκοσμίω, να προστατεύονται παγκοσμίω. Αυτή είναι η βάση και το θεμέλιο της. Η κατάργηση της θανατικής, η ημέρα υπέρ της κατάργησης θανατικής ποινής είναι κάτι που μας θυμίζει ότι υπάρχουν ακόμη χώρες που την εφαρμόζουν και γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας και να τις εντείνουμε κι άλλο. Η αντίθεση, στεναρή αντίθεση της Ένωσης προς τη θανατική ποινή την τοποθετεί στο προπύργιο του αγώνα αυτού και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το πρώτο πολιτικό όργανο που, την εφαρμόζει, που εφαρμόζει αυτόν τον αγώνα. Πρέπει όμως να καταλήξουμε σε μια παγκόσμια απαγόρευσή της, κατάργησή της. Το ΕΛΚ θεωρεί ότι η καταπολέμηση παγκοσμίως της θανατικής είναι μία από τις κυριότερες προτεραιότητες της εξωτερικής μας πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ένωση πρέπει να συνεχίσει να θέτει το θέμα και να υποστηρίζει πρωτοβουλίες που να μπορούν να οδηγήσουν στην παγκόσμια κατάργηση. Θα ήθελα βέβαια επίσης να ζητήσω από την ε, είπα τη εκπρόσωπο την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να μην εγκρίνουν τα χώρι, τις χώρες που δεν έχουν ακόμη εγκρίνει το συναπτώμενο πρωτόκολλο και το πρωτόκολλο 13 στην ε, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να το πράξουν. Η Λευκορωσία είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που εφαρμόζει ακόμη στην πράξη τη θανατική ποινή πρέπει να κάνουμε ό,τι προσπάθεια μπορούμε για να αλλάξει αυτό. Επίσης η Ένωση πρέπει συνεχώς να γνωστοποιεί το πρόβλημα και στις διμερείς της διαπραγματεύσεις και σε διεθνή βήματα. Για να καταλήξω κυρία Πρόεδρε, η Ένωση πρέπει να αποτελέσει έμπνευση προς τον υπόλοιπο κόσμο. Λίγες μέρες μένουν πριν την, τον εορτασμό και γι' αυτό είναι η καταλληλότερη στιγμή να το ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος της Προοδευτικής Συμμαχίας, ο κύριος η κυρία Γκόμες για τρία λεπτά. Η, Μπιλορου... η Λευκορωσία, η Κίνα, το Ιράν, η Σαουδική Αραβία και το Σουδάν τι έχουν ε, κοινό όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Αυτές οι χώρες εξακολουθούν να έχουν κοινή μια πρωτόγονη και φρικτή πρακτική, την θανατική ποινή. Ορισμένα κράτη χρησιμοποιούν αυτή την ε, βάρβαρη μέθοδο ε, μυστικά, χωρίς να μπαίνουν στις στατιστικές. Κίνα, Μαλαισία, Αίγυπτος, Βιετνάμ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκλείσει τη θενατική ποινή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από την Λετωνία να καταργήσει για αυτή τη δυνατότητα που προβλέπεται από το Σύνταγμα μόνο για πάρα πολύ σοβαρά εγκλήματα. Ε, έχουν, ε, γίνονται συσκέψεις κορυφής, πολυμερείς, διμερεί, διαπραγματεύσεις ε, διεθνών οργανισμών, επίσημες επισκέψεις ή στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής αλλά και της ε, οικονομικής συνεργασίας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να τονίζει το θέμα του καθολικού μορατόριου του Γενικής Συνέλευσης. Είπατε εκπρόσωπος η Κάθρινα Αστών θα πρέπει να μέσω της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης να προωθήσει την δράση για την καταπολέμηση της θανατικής ποινής. Υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος. Υπάρχουν ακόμα 54 ε, κράτη-μέλη τα οποία κατήργησαν είτε μέσω του νόμου είτε μέσω της πρακτικής τους ε, την θανατική ποινή πράγμα που είναι πολύ θετικό. Θα πρέπει να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην καθολική κατάργηση της θανατικής ποινής. Κάνω μια έκκληση στην ύπατη εκπρόσωπο επίσης για να προωθήσει το σύστημα αναγνώρισης όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο σε οποιαδήποτε χώρα της Ένωσης και να κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις της για να τους σώσει από αυτή την κατάσταση. Όσον αφορά την εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελπίζει πως θα γίνει σύντομα η αναθεώρηση των ευρωπαϊκών οδηγιών για την θανατική ποινή που προβλέπεται για τον επόμενο χρόνο. Η Ένωση θα πρέπει μόνο να εγγυηθεί την υποχρέωσή της σύμφωνα με το χάρτη των διεθνών ε, συμφωνιών. Άρα λοιπόν ε, ότι δεν υπάρχει καν ο κίνδυνος να βρεθεί κανείς ε, κατηγορούμενος και με την δυνατότητα επιβολή ανετική ποινή, να μην μπορεί κανένα να τεθεί σε τέτοιο κίνδυνο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι σαφέ σε αυτό το ψήφισμα να εκφράζει την αποστροφή του για αυτές τις ε, βίες μορφές ε, ε, τιμωρίας όπως είναι ο λιθοβολισμός. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι, άντρες και γυναίκες που, που βλέπουν τους διαδρόμους του θανάτου στις χώρες τους και βλέπουν με συμπάθεια τους συνανθρώπους τους. Γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας για να τους βοηθήσουμε και να τους σώσουμε. Σας ευχαριστώ εξ ονόματος της Άλντε, ο κύριος Σάκη για δύο λεπτά. Η κυρία Σάκη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Σασέλ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να θεωρήσει προτεραιότητα την καταπολέμηση της θεματικής ποινής παγκοσμίω σε, σε με υποψήφιες χώρες ή τρίτες χώρες όπως το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχώς τονίζουμε τη σημασία που έχει η κατάργηση αυτής της απάνθρωπης ποινή. Δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτρεπτική η θανατική ποινή για την αύξηση της εγκληματικότητας. Δεν ζητούμε βέβαια ατιμορρησία γενικά για τα εγκλήματα, αλλά μόνο Είμαστε κατά της θανατικής ποινής στεναρα. Θεωρούμε ότι πρέπει να καταπολεμάται το έγκλημα διεθνώ πάντοτε όμως με δίκαιε δίκες. Συχνά δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν καθορίσει ότι τα εγκλήματα που αφορούν τα ναρκωτικά δεν είναι από τα σοβαρότερα ούτως ή άλλως. Επίσης έχουν ζητήσει τα Ηνωμένα Έθνη μορατόριου για την θανατική ποινή. Βέβαια, αφού είναι και το Ιράν μέλος της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των γυναικών, η κατάσταση γίνεται κομική. Σήμερα, εδώ στις Βρυξέλλες, διοργανώνεται η, διάσκεψη, η πολιτιστική διάσκεψη Ένωσης Κίνας. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι η Κίνα έχει από τον μεγαλύτερους αριθμούς επιβολής της θανατικής πηγής, πίνης και στη δεύτερη θέση για την εκτέλεση νέων και εφήβων έχει το Ιράν. Το να μιλάμε για πολιτιστικές σχέσεις σημαίνει ότι μιλάμε για βασικές ελευθερίες και πολλοί θανατώνονται ακριβώς γιατί εκφράζουν την πολιτιστική τους ελευθερία. Πρέπει όσο το δυνατόν γρηγορότερα να καταργηθεί παγκοσμίω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τους πράσινους ο κύριος Λοκμπίλερ για δυόμιση λεπτά. Η κυρία Λόκμπιλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκδίδεται κάθε χρόνο κατά της εθελοντικής ποινής για το πόσο μπορούμε να καταφέρουμε υπέρ της κατάρριξη. Ναι, πολλές είναι ακόμη οι περιπτώσεις των θανατικών ποινών που εκτελούνται, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα και ο εκπρόσωπος της ΥΠΑ της εκπροσώπου και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, θα πρέπει να λησμολούμε ότι ο παγκόσμιος αγώνας, στην, ε, ο, ο αγώνας μάλλον σε ολόκληρο τον κόσμο, ο, κατά της στρατικής ποινής ε, είναι ένας επιτυχημένος αγώνας. Είναι ήδη πολλά τα κράτη τα οποία έχουν καταργήσει επίσημα τη θανατική ποινή από την νομοθεσία τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωταγωνιστής των αγώνων αυτών. Τον, ε, το θέμα της θανατικής ποινής το εισάγει σε κάθε διμερή σχέση και δεν πρέπει πιστεύω να να μειώσουμε αυτή την πίεση που ασκούμε στα άλλα κράτη. Και πρέπει να προχωρούμε κατά τρόπο πιο στοχευμένο, διότι βέβαια δεν έχει τι ίδιε δομέ και τι ίδιε δυνατότητε κάθε κράτο και κάθε ε, κυβέρνηση. Και θα πρέπει να αξιοποιούμε διαφορετικέ στρατηγικέ. Άλλο φερρυπίν ε, σύστημα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην ε, Ιαπωνία, όπου σε μία ε, ε, προεκλογική εκστρατεία μόνο μπορεί να επικαλέσει ένα υποψήφιο στο ζήτημα τη θανατική ποινή και άλλοι απέναντι στη Ρωσία ή, την, το Ιράν. Επίση, πάνω απ' όλα θα πρέπει να επιμείνουμε ώστε να μην εκτελούνται τουλάχιστον ανήλικοι ή ε, άτομα με πνευματικά περιορισμένε δυνατότητε. Ή επί παραδείγματι να μην εκτελούνται θανατικές ποινές για πτέσματα τύπου περιουσιακού όπως βλέπουμε να γίνεται ακόμη στην Κίνα με στόχο τελικό βέβαια την τελική και ολοκληρωτική κατάργηση της θανατικής ποινής από, από κάθε κράτος του κόσμου. Σε αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να επαναπαυθούμε στις δάφνες μας, αλλά πάντως δεν θα πρέπει να κρίνουμε και αυτό, σε αυτό θα επιμείνω, με διαφορετικά μέτρα και σταθμά τα κράτη εκείνα τα οποία ακόμη διατηρούν τη θενατική ποινή ανάλογα με τις σχέσει που έχουν μαζί του. Το φετινό μα ψήφισμα για την κατάρρηση θενατική ποινή ιδιαίτερα εστιάζεται στι ΗΠΑ και ιδιαίτερα υποδειγματικά θα ήθελα να αναφέρω μία περίπτωση τη Μούμια Αμπουτζαμάλ, η οποία έμεινε επί 20 χρόνια, μένει επί 20 χρόνια θανατοπινίτησα. Είναι μια Αφροαμερικανίδα η οποια εμεινε επι 20 χρονια μενει επι 20 χρονια θενατοποινητησα ειναι μια αφροαμερικανιδα η οποια είχε δραστηριοποιηθεί στην δημοσιογραφία την μαχόμενη, τη ριζοσπαστική και μαχόμενη δημοσιογραφία και φαίνεται ότι η καταδίκη της οφείλεται σε κάποια ε, τυπικά ελαττώματα της δίκης. Γι' αυτό πρέπει να αγωνιστούμε όλοι, ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να συναντηθεί η ευκαιρία για μια δίκαιη δίκη. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, ο κύριος Κάριμ. Για ένα λεπτό. Mm-hmm. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ενώ μιλώ εξ ονόματο τη ομάδα ε, των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, τα σχόλιά μου βασίζονται στι αποκλειστικά στι προσωπικέ μου πεπιθήσει. Καλωσορίζω τη σημερινή συζήτηση, γιατί αποτελεί μια απόδειξη τη αφοσίωσή μα ε, στι βασικέ αξίε τη Ένωση. Πέρσι, τουλάχιστον 714 άνθρωποι εκτελέστηκαν από κράτη αυτό χωρίς την Κίνα, γιατί εκείνοι δεν έχουν διαφάνεια για το θέμα. Πολλά κράτη που ακόμα ισχύει η θανατική ποινή ως ε, εργαλείο τιμωρίας δεν έχουν το μηχανισμό ώστε να δώσουν δίκαιη δίκη για αυτούς που κατηγορούν για ε, εγκλήματα ε, που αξίζουν τη θανατική ποινή. Διατηρούν έτσι τη δυνατότητα να μην πραγματοποιήσουν τη θανατική ποινή Πράγμα το οποίο είναι ε, δεν είναι τόσο δραματικό όσο αρχικά μπορεί κανείς να φανταστεί. Τα στοιχεία ωστόσο που σας έδωσα δεν αναφέρουν τον κόσμο που περιμένει καταδικασμένος και περιμένει να δει ποια θα είναι η μοίρα του. Πολλοί είναι αθώοι και δεν έχουν μπορέσει καν να δικαστούν δίκαια. Ενώ κάνουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση, είναι μια προσωπική συζήτηση, δεν αφορά μόνο εκείνους που αντιμετωπίζουν την καταδίκη σε θανατική ποινή, αλλά και ένα σωρό κόσμο που επηρεάζεται από αυτό, όπως οι οικογένειέ του και τόσος κόσμος στην κοινωνία, απλά και μόνο γιατί οι άνθρωποι περιμένουν να εκτελεστούν χωρίς καμία δυνατότητα για δίκαιη δίκη. Θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και σε αυτές τις περιπτώσεις. Grazie. ευχαριστώ. Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς και Βόρειας Πράσινης Αριστεράς, ε, ο κύριος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η πρόταση ψηφίσματος που εξετάζουμε σήμερα καθορίζει τους όρους της αντίθεσής μας προς τη θανατική ποινή. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για κανένα κράτος ώστε εν ψυχρό <coughs> να αποφασίζει τη θανάτωση πολιτών του και η θανατική ποινή είναι και η ίδια ένα έγκλημα. Πολύ συχνά και κάτι ακόμα παραπάνω. γιατί πρόκειται και για βασανιστήριο όσο κανείς αναμένει την εκτέλεσή του. Χρησιμοποιείται προς εκφοβισμό ορισμένων καταπιεσμένων πληθυσμών όπως το Ιράν. Είναι λοιπόν και τρομοκρατία η θανατική ποινή. Ο δημοσιογράφος Μούμια Μποτζαμάλ που αποτελούσε όπως λέγανε την φωνή των αφώνων είναι ένα σαφές σύμβολο. Κατηγορήθηκε για τη δολοφονία ενός αστυνομικού και καταδικάστηκε σε θάνατο. Και δεκαετίες ανέμενε μετά από διαδικασίες δικαστικές όπου χαρακτηρίζονταν από κατάφορο ρατσισμό. Είναι λοιπόν ένα από τα πιο σημαντικά παραδείγματα που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στον αγώνα μας. Εφόσον μάλιστα οι εκπρόσωποι, όταν μάλιστα οι εκπρόσωποι της Ένωσης θα συναντηθούν την επόμενη φορά με Αμερικανούς αξιωματούχους ή τον ίδιο τον πρόεδρο. Και το παράδειγμα αυτό που σας ανέφερα είναι σημαντικό γιατί προέρχεται ακριβώς από τις Ηνωμένε Πολιτείε που είναι ο κυριότερος σύμμαχος της Ένωσης. Στην καταπολέμηση λοιπόν, για την, στον πόλεμο για την κατάργηση της θανατικής ποινή, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά αλλά μόνο ένα μέτρο και ένα σταθμό δηλαδή όχι στη θανατική ποινή. Όχι. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μπιτζότο. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει η Ευρώπη να πιέσει όσο μπορεί για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Πέρα από τις δηλώσεις των αρχών πρέπει η Ένωση να εφαρμόσει συγκεκριμένα εργαλεία, αυτά που διαθέτει. Πολλές τρίτες χώρες εφαρμόζουν τη θανατική ποινή με βαρβαρότατο τρόπο και παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση συνάπτει εμπορικές συμφωνίες μαζί τους. Πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε προς τις χώρες αυτές ώστε να σεβαστούν και αυτές τα ελάχιστα πρότυπα για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πράγμα το οποίο δυστυχώς δεν συμβαίνει. Καμιά φορά η Ευρώπη κλείνει τα μάτια. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε με την Κίνα, την Ιεμένη, το Πακιστάν και με τέτοιε χώρε να έχουμε εμπορικέ συμφωνίε και να μην μιλάμε για τη θανατική ποινή. Αυτά είναι βασικά στοιχεία τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να καταργηθεί η θανατική ποινή, διότι δυστυχώ μέχρι τώρα, όπω είπα, η Ευρώπη δεν το έχει πράξει μέχρι τώρα. Σα ευχαριστώ από του μη εγγεγραμμένου. Ο κύριο Γκόρνη για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, για την 8η ε, Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής θα ήθελα να μιλήσω, να εκφράσω τις σκέψεις μου για όλους αυτούς των οποίων θανατική ποινή δεν εορτάζουμε. Την Αν Μουζέλ που εκτελέστηκε πριν από μια εβδομάδα περίπου με Κατσαβίδη από έναν ε, υπότροπο εγκληματία για ε, παιδιά, για ένα τετράχρονο που δολοφονήθηκε, για έναν γέροντα στην περιοχή μου που δολοφονήθηκε από υπότροπο για τα 400 εκατομμύρια παιδιά που αγέννητα ακόμα δολοφονούμε στην κοιλιά της μητέρας σου κάθε χρόνο, για τη Μαρή Κριστίν, τη Μέρη Κρετμέλ ε, και άλλους που το μόνο τους σφάλμα ήταν να βρεθούν στο δρόμο ενός αποτρόπαιου εγκληματία που απελευθέρωσαν οι αρχές. Για όλα τα θύματα του Ντιτρού, του Ευράρ, του Φουρνιρέ. Όλου, όλα αυτά τα θύματα που κι αν ακόμα δεν έχασαν τη ζωή τους ή την είδαν να καταστρέφεται οριστικά. Για όλα τα θύματα της Μαδρίτης, του Λονδίνου, τα θύματα της τυφλής Διβίας, για τα οποία δεν ε, ορίζουμε ε, παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματά τους. Όμως, παγκόσμια ημέρα για, τα, για τους θύτες τους, για τους δημίους τους, ορίζουμε και εορτάζουμε. Ζητούμε να καταργηθεί η θανατική ποινή αυτών των εγκληματιών. Θανατική ποινή που μερικές φορές είναι ο μόνος δρόμος λύτρωσης για τα θύματα τους. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Και τώρα Δίνουμε το λόγο και πάλι στο Συμβούλιο και μετά θα παρακαλώ. Και ω εκ τούτου παρακαλώ τον κύριο Σαστέρ να λέει το λόγο. Πρόεδρε. Ξέρω ότι είμαι κυρίε και κύριοι βουλευτέ. Δεν μου μένει παρά να σα ευχαριστήσω για τι παρεμβάσει σα. Βλέπω ότι σχεδόν ομόφωνα μα υποστηρίζετε στι πρωτοβουλίε και τι δράσει μα. Άρα συμφωνούμε ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδώσει ιδιαίτερη σημασία στη δράση αυτή για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Όπως ανέφερα και νωρίτερα, η είπατε εκπρόσωπος, κυρία Άστον, έχει καταστήσει το στόχο αυτό προσωπική της προτεραιότητα και επιθυμούμε διακαώς να καταστεί ο στόχος αυτός επιτυχής, όπως άλλωστε υπογραμμίσαμε και στην 65η Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών, και με ένα ψήφισμα που θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο το κίνημα για ένα παγκόσμιο μορατόριο της θανατικής ποινή. Διότι θεωρούμε ω θεμελιώδη αρχή ότι είναι απαραίτητο να καταργηθεί θανατική ποινή ως ένδειξη σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Και γι' αυτό εν πάση περιπτώσει για κάθε αδίκημα και για κάθε περίσταση σώμεθα υπέρ της κατάργησης της εσχάτης των ποινών. Είπαμε και πριν ότι δεν υπάρχει περιθώριο αυταρέσκειας, επανάπαυσης και ως εκ τούτου αξιοποιούμε κάθε μέσο που έχουμε στη θέση μας για την επιτεύξη του στόχου αυτού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να σας ανακοινώσω ότι έχω λάβει πέντε προτάσεις ψηφίσματος. Ε, σε σχέση με αυτό το θέμα. Τώρα ολοκληρώνεται η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Ora l'ordine del giorno reca l'interrogazione